Herzlichen Dank. Hier wird jeder zu Wort kommen. Jetzt aber zunächst der Kollege Berlinguer. Bitte. Sì, io mi unisco alle considerazioni del nostro Presidente circa il ringraziamento alla Vicepresidente e Commissaria signora Reding e al modo in cui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 ganz, ganz wichtiges Element für zukünftige Rechtsentwicklung in Europa. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Lichtenberger. Frau Kollegin Morvay, bitte. Thank you very much. We have in our hands this beautiful new booklet on the EU Justice Scoreboard. And on page three, we can read, let me quote,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 30, und zwar unter Verschiedenes, das Thema Implementing Enhanced Cooperation in the Area of Financial Transaction Tax. Das Wort hat Frau Kollegin Regner. Bitte. Dankeschön. Η κυρία regner Ρέγνερ, σας ευχαριστώ πολύ. Η φορολογία επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μακρά ιστορία πίσω τους. Ε, εδώ και αρκετά χρόνια, κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, ε, το Κοινοβούλιο έχει επαναλάβει την ανάγκη ύπαρξη ενός ε, τέτοιου φόρου. Και σε ψηφίσματα το έχουμε εκφράσει αυτό. Από την Κομισιόν. Όμως δεν είχαμε λάβει σχετική πρόταση. Τώρα έχουμε καταλήξει στην διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας και από φέτος τον Φεβρουάριο έχουμε την πρόταση της Κομισιόν ε, που θα πρέπει να αποφασιστεί από 11 κράτη-μέλη και γι' αυτό βρίσκεται και στη μέση διάταξη. Η διαδικασία που έχει επιλογή είναι μία όχι πολύ συνηθισμένη και θα ήθελα γι' αυτό να την ε, περιγράψω σύντομα. Είναι, όπως είπα, πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Η ΕΚΟΝ ε, πιέζει, θέλει τον Μάιο να ψηφίσουμε στην Επιτροπή το θέμα αυτό και γι' αυτό έχουμε αποφασίσει ε, μία μη συνηθισμένη διαδικασία. Ε, να μην στείλουμε υπομορφή επιστολής την γνωμοδότηση, αλλά να ψηφίσουμε τις τροπο, τροπολογίες αύριο ώστε να έχουμε κάπως πιο νομικά έγκυρη μορφή. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν αύριο να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Στην ε, τελευταία ολομέλεια του ε, Στρασβούργου είχαμε μία ε, συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές και προσπάθησα να συμπεριλάβω υπόψη μου όσο γίνεται περισσότερα από αυτά που άκουσα. Η κυρία Λίχτενμπεργκερ έχει ε, τηρήσει την ε, προθεσμία ε, και θα υπάρξουν και προφορικές τροπολογίες. Πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ στο περιεχόμενο, διότι η πρόταση της Κομισιόν γενικά βρίσκει την συμφωνία μας, πιστεύω ότι είναι καλή, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στα εξής. Η Κομισιόν διασαφηνίζει ότι τα παράγωγα καλύπτονται από τον φόρο αυτόν και για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό ε, να μην αποδυναμωθεί αυτό και γι' αυτό ιδιαίτερα θέλουμε να αναφέρουμε τα CFD, διότι η ίδια η Κομισιόν ε, πριν κάποιες ε, εβδομάδες ε, προειδοποίησε τους ε, μικρούς ε, καταθέτες κατά αυτών των CFD, διότι μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες απώλειες και ζημίες. Και θα ήθελα να πω ότι ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από εισαγωγή του, των χρηματοοικονομικών τελών εξαφανίστηκαν τα προϊόντα αυτά το όλο θέμα αυτό σχετίζεται και με τον, την καταπολέμηση των φορολογικών ε, παραδείσων. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα σφαιρικά. Ε, δεν θέλουμε λοιπόν να καταπολεμήσουμε μόνο την φοροδιαφυγή, αλλά και την ε, ε, συνειδητή φοροαποφυγή και γι' αυτό υπάρχει μια τροπολογία η οποία περιορίζεται στην φόρο ε, διαφυγή, αλλά θέλουμε εμείς να αναφέρουμε και την συνειδητή φόρο αποφυγή. Και τέλος ε, θα ήθελα να αναφέρω, διότι είναι μια πληροφορία που ίσως να έχετε λάβει, ίσως όχι, ότι από ανακοινοθέντα τύπου μαθαίνουμε ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ε, ε, έχει πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, λόγω της ενισχυμένης συνεργασίας. Ιδιαίτερα δεν, την, δεν της αρέσει το πεδίο εφαρμογής του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και πιστεύουμε ότι πρόκειται για ε, μια προσπάθεια για να καθυστερήσει το όλο θέμα και πιστεύω ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την όλη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ζητάει κανείς το λόγο. Μια παρατήρηση να κάνω ότι αυτή η στρατηγική ε, είχε αποτύχει και με τα διπλώματα έβρεση τεχνίας. Η διαδικασία είναι μια διαδικασία σου generis. Ε, φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχουν αντιρρήσεις. Ε, άλλωστε όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούσαν, ε, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Κλείνουμε λοιπόν το γενικό κομμάτι της συνεδρίασης και προχωράμε στην συνεδρίαση και των θυρών. Παρακαλώ να κλείσουμε την ε, την ε, μετάδοση από το ίντερνετ ε, και διάλειμμα δύο λεπτά. Παρακαλώ να καταλήψουν την αίθουσα όσοι δεν πρέπει να είναι παρόντες.